Θα ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία σε λίγα δευτερόλεπτα. Χρειάζεται να έχετε την κάρτα σας όλοι και να μας ενημερώσετε αν δεν την έχετε. Ευχαριστώ. Άννα Μαρία, έρχεται. Προς τους συναδέλφους ε, που δεν ήταν εδώ σήμερα το πρωί, καλώς ορίσατε, καλώς επιστρέψατε από τις καλοκαιρινές διακοπές. Όποιος δεν έχει την κάρτα ψηφοφορίας μπορεί να με ενημερώσει τώρα. Έχουμε ήδη ένα μέλος που δεν την έχει και βρίσκεται καθοδόν. Κανείς άλλος. Ωραία λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουν όλες τις κάρτες. Okay, colleagues, everyone, please take Συναδέλφοι, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία για το Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό έτο 2017. Έχουμε δύο λίστε ψηφοφορία, μία για την γνωμοδότηση και μία για τι ε, τροπολογίε του ε, προπολογισμού. Οπότε ξεκινάμε με την ε, λίστα ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση. Και ξεκινάμε με την έγκριση της νομοδότησης τη κυρίας Μακοβέη. Θα δούμε όλες τις τροπολογίες και μετά θα περάσουμε στις 64 ε, ε, τροπολογίες του προπολογισμού που περιλαμβάνουν και πολλά ε, σχέδια. Η κυρία Μακοβέη θέλει να πει δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες ε, του προϋπολογισμού για τον προϋπολογισμό του 2017 και την ογνωμοδότηση της ΛΥΜΠΕ για τον προϋπολογισμό αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το έργο τους, για τη συμβολή τους, ε, ώστε να ολοκληρωθεί το έγγραφο. Ε, ελπίζω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας να δείξει στους Ευρωπαίους πολίτες ότι είμαστε υπεύθυνοι και ότι έχουμε πάρει σοβαρά τις προτεραιότητε του προπολογισμού για το 2017. Πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, μην ξεχνάμε τα σημαντικά. Η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών αποτελεί προτεραιότητα για μα και αυτό εμεί πρέπει να το δείξουμε ορίζοντα τι σωστέ προτεραιότητε στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, τα χρήματα των πολιτών πρέπει να δαπανηθούν ε, στις σημαντικές προτεραιότητες και τα σημαντικά προγράμματα που αφορούν σοβαρά θέματα. Πρέπει να σεβαστούμε το έργο τους και τη συμβολή τους στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Ευχαριστούμε. Ας προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, κάτι λάθος έχει γίνει με αυτό το μηχάνημα. Δεν φαίνεται να λειτουργεί. Ας προσπαθήσουμε ξανά δεν λειτουργεί. Σίλια, θέλετε να πάτε σε μια άλλη θέση. Θέλετε να πάτε σε ένα άλλο μηχάνημα, να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Αλλάξτε απλά θέση και... Thank you for that. Thank you for that helpful... Ευχαριστούμε για την ε, χρήσιμη πρόταση στο μας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, οπότε θα συμπεριλαμβάνουμε ό,τι κάνατε στα πρακτικά. Λειτουργεί. Δύο μηχανήματα δεν λειτουργούν. Τι είναι το άλντε πλήτη αυτή η κατάσταση. Δουλεύει. Ωραία, λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Θα αναφέρουμε την ψήφο σας στα πρακτικά. Λοιπόν, συμβαστική 2, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρινέται ε, τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται τροπολογία 18. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 19. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 20. Άρχεται ψηφοφορία. Κλείνει. Απορρίπτεται 21. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 22. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 24 άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 27 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 32. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 33. Ε, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 35. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Τμήμα 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 4 τμήμα 2, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 45, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 46, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48, άρχεται ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται 55 άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 56 άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 57 άρχεται ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. 58 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. εγκρίνεται με ένα σφάλμα από το ΕΛΚΑ 51. Τμήμα 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 61, έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 62, η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 63, η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 64 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 65 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 66 άρχεται η ψηφοφορία. πέρας απορρίπτεται και περνάμε στην τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρινέται 43 υπέρ 6 κατά 3 εποχές περνάμε τώρα στις τροπολογίες του προπολογισμού And we start, colleagues, with the oral budgetary amendment. Προφορική τροπολογία του ΕΛΚ, Σοσιαλιστών, ΑΛΔΕ και ΓΟΕ για να επανέλθει η δημοσιονομική θέση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Κομισιόν, συγγνώμη. Η είναι κατά ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας της ίδιας αυτής της ψηφοφορίας γίνεται δεκτή η τροπολογία. Hey, colleagues, um, now the budgetary amendments, Libby 5. Τροπολογίες 54-95. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 54-72. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 54-69. Άρχεται. Δεν την κλείσαμε καλά την προηγούμενη ψηφοφορία. Μια στιγμή να ξαναπέρα ψηφίσουμε την 54-92. Γιατί απερίφθη Μπορούμε να κάνουμε μια λέγη. λοιπον 5492. 5492, 54 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 54-69. Άρχεται. Περαίνεται. Απορρίπτεται. 54-70. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 54-50 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 54-71 άρχεται. Πέρασε. απορριπτεται Απορρίπτεται. 54-94 άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Αρχή ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 54-51. Άρχεται. Πέρας απολυτωται 54 54-76. Αρχίζει. Τελειώνει. απολυτωται 55 55-03. Άρχεται. Πέρασε παιχτη 54 54-77 αρχίζει. Τέλος. απολυπτεται 54 54-52 έναρξη. Τέλευση. Απολύπτεται. 54-78 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται 54-79 έναρξη. Τέλος. Απορρίπτεται. 54-53 έναρξη. Τέλος. Απορρίπτεται. 54-62. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 54-80. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 54-74. Άρχεται. Πέρας. Απολύπτεται. 54-54. Αρχίζει. τελος Απολύπτωται Απορρίπτεται. 54-63. Αρχίζει. τελος Απολύπτωται Απορρίπτεται. 54-75. Αρχίζει. Τέλος. Απολύπτεται. έναρξη. Τέλος. Απολύπτεται. έναρξη. Τέλος. Απορρίπτεται. 54-82. Άρχεται. Πέρας. Απέριπτε. 54-86. Έναρξη. Τέλος. Απορρίφθηκε. 54-57. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 54-88. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 54-89. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 54-98. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 54-87 άρχεται. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 54-65 άρχεται. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 54-59 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 54-60. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 54-68. Άρχεται. Πέρας. Απολύτωται. 54-56. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πενήντα τέσσερα, ογδόντα Έναρξη. Τέλος. Απορρίφθηκε. 54-67. Έναρξη. περασε απορριφθηκε Απορρίφθηκε. 54-55. Έναρξη. Τέλος. Εγκρίνεται. 54-85 άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 5491 άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 5458 άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 5490 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 55 55-06. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 5 5509. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 5461. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 5508. Αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. 5500. Αρχίζει. Πέρας. Απορρίπτεται. 55-13. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. 55-02. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 55-04. Άρχεται. Τέλος, εγκρίνεται. 54-99. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίθηκε. 55-01. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 5-5-10. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Υπάρχει τελική ψηφοφορία. Έχουμε τελειώσει. Τελειώσαμε και συγχαρητήρια στην κυρία Μακοβέη, την εισηγητρία μας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για την παρουσία σας τέρμα ο χρόνος ψηφοφοριών. Nice to see you, though. Colleagues, I'm just going to make a quick announcement about timing. Συνάδελφοι, θα κάνω μια σύντομη ανακοίνωση για τα προγράμματά μας όσοι επανέρχεστε από τα σημεία 11 και 12. Τα σημεία 11 και 12. Τα 11 και 12 λοιπόν θα τα δούμε στις, 6, ε, στις 4 και μισή, μια ώρα διάλειμμα δηλαδή, στις 16 και 30 τέσσερις και μισή, γιατί τελειώσαμε πολύ νωρίτερα τις ψηφοφορίες μας από ό,τι περιμέναμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν τα σημεία 11 και 12 στις 4 και μισή. Διάλειμμα για μια ώρα, γιατί είμαστε τόσο αποτελεσματικοί. Κουρασμένοι είμαστε. Ζήτω συγγνώμη που σας κάνω να περιμένετε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Dear Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι ο χρόνος πέρασε και μπορούμε να επανέλθουμε. Καλώς ήλθατε και πάλι στις 4.30 στην αίθουσά μας. Ευχαριστώ που προσαρμοστήκατε στο χρονοδιάγραμμα. Τελειώσαμε λίγο νωρίτερα τις ψηφοφορίες και τώρα και ο κύριος Δίας Μέρα είναι εδώ παρόν, ο εισηγητής μας. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 11 της τη διάταξης, που είναι η ανακοίνωση της Κομισιόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την κατάσταση των πραγμάτων και την ε, πορεία προς το μέλλον για την κατάσταση μη αμοιβαιότητας με τις τρίτε χώρες στον τομέα της πολιτικής προξενικών θεωρήσεων. Συνέχεια της ανακοίνωση της 12 η Απριλίου θα έχουμε μια παρουσίαση από τον κύριο Ολιβιέ Ονίδη, γενικό, αναπληρωτή γενικό διευθυντή τη DG και ως εισαγωγή, ειδού ο κύριος Ονίδης, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω ότι στις 13 Ιουνίου, Ιουλίου, στις 13 ε, Ιουλίου η Κομισιόν παρουσίασε μια περαιτέρω ανακοίνωση σε σχέση με το να αντιμετωπιστούν καταστάσεις μη αμοιβαιότητας για τα θέματα προξενικό θεωρήσεων. Κάποιοι πολίτε ορισμένων κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται βίζα για να πάνε στι ΗΠΑ και στον Καναδά. Και ενώ οι Καναδοί και οι Αμερικάνοι δεν χρειάζονται βίζα για να μπουν στην περιοχή του Σέγγεν. Αυτό λοιπόν είναι συνέχεια στην ανακοίνωση 10 Απριλίου που συζητήσαμε στι 20 Απριλίου. Στη συνέχεια <clears throat> και επί τη βάση τη απόφαση των συντονιστών τη Επιτροπή μα στι 10 Μαου 10 Ιουνίου έγραψε στον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο τονίζοντας ότι κατά τη δική μας άποψη η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να εγκρίνει μια κατεξουδότηση πράξη βάσει του κανονισμού του 2001 που να ε, αναστείλει προσωρινά την εξαίρεση από την ε, ανάγκη βίζας για κατοίκους τριτών χωρών. Στη συνέχεια η Κομισιόν παρουσίασε μια περαιτέρω ανακοίνωση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ολίβιε Ονίδη για την παρουσίασή του και μετά στα μέλη της Επιτροπής ξεκινώντας με τον κύριο Διασδέ, Μέρα, ο οποίος είναι ο συγητής μας. Έχετε το λόγο κύριε Κονίδη. Παρακαλώ. Περιμένουμε να ακούσουμε τις εξηγήσεις. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ που αφιερώσετε λίγο χρόνο για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και στο τέλος μιας πολύ άσχολης ημέρας. Είπατε ήδη αρκετά και συνοψίσατε πολύ σωστά ότι μετά από την επιστολή σας στην Κομισιόν στις 7 Ιουνίου αποφάσισαν οι Επίτροποι να μην χρησιμοποιήσουν κατεξουδότηση πράξη στην παρούσα φάση δεδομένων κάποιων σημαντικών ε, γεγονότων που έλαβαν χώρα τόσο με τις ΗΠΑ αλλά και με τον Καναδά. δεδομένης της πολιτικής σπουδαιότητας του ζητήματος αυτού έχουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε τακτικά όλα τα θεσμικά όργανα οπότε αποφασίστηκε να εκδοθεί μια νέα ανακοίνωση μετά από αυτήν του περασμένου Απριλίου στις 13 Ιουλίου Δύο σημεία πρέπει να σημειώσουμε κατά βάση όπως περιγράφεται ε, λεπτομερώς στην ανακοίνωση πρώτον το Ιόνσο, ότι το Μπρουνέι έχει άρει όλες τις απαιτήσεις ε, ε, προξενικών θεωρήσεων για όλους τους Κροάτες πολίτες, γεγονός που σημαίνει ότι το Μπρουνέι πλέον δεν ε, παρουσιάζει πλέον πρόβλημα με αμοιβαιότητα όσον αφορά τις θεωρήσεις και μετά όσον αφορά την κατάσταση με τον Καναδά και τη ΣΥΠΑ παρέχεται μια λεπτομερή εικόνα στα δύο που βρίσκονται οι συνομιλίες με αυτούς τους δύο σημαντικούς εταίρους όσον αφορά τον Καναδά ε, που είναι η πλέον υποσχόμενη πλευρά ε, ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος ε, είχε μια αναλυτική συζήτηση με τον Καναδό ομολογό του, τον Υπουργό Μακάλλαν στις 11 Ιουλίου Αποφασίστηκε μια ιδιαίτερη σύνθεση για τις συνομιλίες αυτές, διότι αποφασίστηκε τόσο από την καναδική πλευρά όσο και από τη δική μας πλευρά ότι καλό θα ήταν να συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις ε, ο Ρουμάνος και ο Βούλγαρος ε, ε, υπουργός ώστε να συζητηθούν όλα τα ζητήματα. Η συζήτηση αυτή οδήγησε σε μια πολύ ικανοποιητική δήλωση που συνοψίζει πιστεύω το πνεύμα που επικράτησε στη συνάντηση. Μια ειλικρινής κατανόηση ότι ο Καναδάς πρέπει να προβεί σε άρση των όσων περιορισμών απομένουν όσον αφορά τις θεωρήσεις και καταρτίστηκε και ένας λεπτομερής οδικός χάρτης. Η δήλωση αυτή ακολουθήθηκε αμέσως από κάποιες ε, τεχνικές αποστολές. Καναδοί αξιωματούχοι ουσιαστικά μετέβησαν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία ε, για να διεξάγουν λεπτομερή συζητήσεις και με τις δύο πλευρές ε, ώστε να διευκρινιστούν οποιαδήποτε ερωτήματα απέμεναν αλλά και ώστε να καθισχαστούν, να, να καθισχάσουν η ρωμανική και η βουλγαρική πλευρά τις κρατικές αρχές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κατάχρηση του καθεστώτος της άσκηση των θεωρήσεων. Το επόμενο βήμα θα λάβει χώρα αυτή την Κυριακή. Επειδή το ζήτημα αυτό απασχολεί πολύ σοβαρά το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, στο πλαίσιο του G20 την Κυριακή θα έχει μια συνομιλία με τον Πρωθυπουργό κ. Τριντό και θα θέσει το ζήτημα αυτό. Και ξέρετε πως η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν συνδέσει αυτό το ζήτημα με δύο σημαντικές συμφωνίες ε, με τον Καναδά, την ΣΕΤΑ και τη στρατηγική εταιρική σχέση. και έχοντα υπόψη το επόμενο σημαντικό ραντεβού με τον Καναδά που θα λάβει χώρα στι 27 Οκτωβρίου όπου θα λάβει χώρα η Σύνοδο κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά. Ελπίζουμε λοιπόν ότι οι συζητήσει θα προχωρήσουν με τρόπο τέτοιο που ο Καναδάς τελικά θα επικυρώσει ότι θα υπάρξει αμοιβαιότητα και άρση τη υποχρέωση θεώρηση για Βούλγαρου και Ρουμάνους πολίτε. Το επόμενο βήμα που περιμένουμε άμεσα είναι στις αρχές του φθινοπόρου να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με τους ε, καναδούς ομολόγους μας όσον αφορά τα αποτελέσματα της εξολόγησης που έκαναν αυτοί τόσο κατά τη διάρκεια των ε, τεχνικών αποστολών ε, στη Βουλγαρία όσο και στη Ρουμανία. Όσον αφορά τη ΣΥΠΑ, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Με τη ΣΥΠΑ τα πράγματα είναι πάντα διαφορετικά. Ε, γνωρίζετε πολύ καλά την τρέχουσα κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα ε, ιδιαίτερο σημείο που συχνά υπογραμμίζουν οι Αμερικανοί ομολογοί μας, ε, κυρίως σε επίπεδο διοίκησης, το γεγονός ότι όλο και περισσότερο στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών τίθεται το ερώτημα των παγίδων που ενέχει το σημερινό ε, καθεστώς θεωρήσεων και θέλουν να προχωρήσουν πολύ προσεκτικά ώστε να μην εγκρίνουν κάτι που δεν θα αρέσει και που ενδέχεται να υπονομεύσει ολόκληρο ε, τη διαδικασία και το σύστημα από αμερικανικής πλευράς ε, γίνονται τακτικές συναντήσεις υπάρχει ισχυρή δεσμεύση από την σημερινή κυβέρνηση για πρόοδο όση πρόοδο προλαβαίνει να γίνει μέχρι το τέλος ε, της θητείας της κυβέρνησης αυτής. Ε, για να καταλάβετε χαρακτηριστικά, η επόμενη συνάντηση εξωματούχων, ειδικά για το θέμα αυτό, έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου. Πολύ σύντομα δηλαδή. Ελπίζουμε ότι και οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να καταλήξουν σε αποτελέσματα, κάτι που αναμένουμε εδώ και καιρό. Και φυσικά θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σας ενημερώσουμε, να σας ενημερώνουμε όπως ε, χρειάζεται και δημερώς ε, ώστε να σας ενημερώνουμε τακτικά για τα όσα συμβαίνουν όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Διαδεμέρα. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ευχαριστήσω και τον κύριο Κουνίδη για τα σχόλιά του. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνουμε τη ίδια συζήτηση που κάναμε στις 20 Απριλίου με μεγάλη προσοχή παρακολούθησα αυτά που είπε ο κύριος ο πρόεδρος της Κομισιόν κύριος Γιούγκερ και συμφωνώ πρέπει να πω απόλυτα με την ε, συνθετική εικόνα που μας έφερε ο κύριος Ονίδη για την προβληματική που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τότε στις 20 Απριλίου έλαβε χώρα μια απόλυτη συνένεση για όλες, από όλες τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να ζητηθεί από την Κομισιόν να τηρηθεί ο κανονισμός 539 κάθετος 2001, ο οποίος έχει τροποποιηθεί από τον 1289 του 2003, το οποίο στάθηκα συγητής. Και μία φορά ακόμα θέλω να τονίσω ότι δεν είναι πρόθεσή μου τώρα να υπησέλθω σε μία αξιολόγηση του περιεχομένου αυτής της δεύτερης ανακοίνωσης πληροφοριακού χαρακτήρα της Κομισιόν που έχω ενώπιόν μου και που έχω αναδιφύσει με μεγάλη προσοχή. Η Κομισιόν νομίζω ότι θεραπεύει τους τύπους, αλλά η ερμηνεία που εγώ μπορώ να αντλήσω είναι ότι δεν λέει τίποτα σε σχέση με τον Μπρουνέι, έχει να πει πολλά σε σχέση με τον Καναδά, Νομίζω ότι μάλλον υπάρχουν πολλά πρέπει να πούμε σε σχέση με τον Καναδά και ακόμα περισσότερα για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Στο κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Νομίζω ότι αυτό που ανέφερε ως επιφυλάξεις η Κομισιόν είναι στην πραγματικότητα συγκεκαλυμμένες απειλές από την πλευρά της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που μας λένε με κάποια ερμητική γλώσσα η οποία είναι όμως κατανοήσιμη αυτό που μας λένε είναι προσέξτε με αυτό που θέλετε να κάνετε γιατί θα μπορούσα να διευρύνω την υποχρέωση για τις προξενικές θεωρήσεις σε 23 κρατημέλη, δηλαδή εκτός από τα 5 που έχουν ήδη μια συμφωνία. Αυτό είναι απόλυτα απαράδεκτο. Βλέπουμε λοιπόν ενώπιόν μας Έχουμε ενώπιον μας την άρνηση του Αμερικανικού Κογκρέσου να κωδικοποιήσει την νομοθεσία του. Όλα αυτά είναι μια γλώσσα, μια διατύπωση, η οποία είναι απόλυτα απαράδεκτη. Ενώπιον λοιπόν αυτή της πραγματικότητα, μετά από αυτά τα οποία εξήγησε και ο κύριος Μωράης, ο πρόεδρος της Επιτροπής μας, έχουμε το άρθρο 1.4.F το οποίο λέει ότι μέσα σε ένα διάστημα 24 μηνών μετά από την δημοσίευση της κοινοποίηση, εάν η τρίτη χώρα δεν έχει άρει την υποχρέωση για βίζα, είναι υποχρεωμένη η Κομισιόν να εγκρίνει μια ε, κατεξουσιοδότηση πράξη με την οποία τροποποιείται ο κανονισμός και για 12 μήνες αναστέλλεται η απαλλαγή από προξενική θεώρηση για τους πολίτες της εν λόγω χώρα. Αυτό αφορά τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τον Μπρουνέι αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι υποχρεωτικό από την πλευρά τη Κομισιόν να πράξει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα, κάποιο τέχνασμα με το οποίο μπορεί να αποφύγει η Κομισιόν αυτή την υποχρέωση. Ο κανονισμός 539 περιλάμβανε κάποιες εναλλακτικές ε, λύσεις, αλλά αφού εγκριθεί η κατεξουσιοδότηση πράξη, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Όπως ξέρετε, στις 12 Απριλίου εξέπνευσε αυτή η προθεσμία των 24 μηνών και αυτή ήταν η χρονική στιγμή όταν η Κομισιόν θα είχε, ήταν υποχρεωμένη να παρουσιάσει μια κατεξουσιοδότηση πράξη. Δεν το έκανε αυτό και αντί, γι' αυτό παρουσίασε μια πρώτη ανακοίνωση. Και τώρα έχουμε τη δεύτερη ανακοίνωση της Κομισιόν ζήτησε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να εκφράσουν την άποψή τους. Μα το κάνουμε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά η Κομισιόν στην ε, κάπως λιθαργική της στάση μας είπε ότι πρέπει να εγκριθεί αυτό από την Ολομέλεια. Μα δεν είναι η εκτελεστική επιτροπή που θα πει στο Κοινοβούλιο πώς θα εγκρίνει ένα νομοθέτημα μέσω της Ολομέλειας, της απόφασης μιας επιτροπής ή μιας επιστολής του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου. Υπήρξε μια σαφής θέση του Κοινοβουλίου η οποία υπηρξε μια σαφη θεση του απερίφραστη και η οποία υποστηρίζεται από όλε τι πολιτικέ ομάδε και δεν χωρεί καμία απολύτω αμφιβολία για τη θέση του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει λοιπόν τη θέση του. Δεν θέλω να επισέλθω στο αν το έκανε το Συμβουλίο, όχι, αλλά το Κοινοβούλιο το έπραξε με απόλυτη σαφήνεια. Ο πρόεδρος Μωράζης στις 7 Ιουνίου απέστειλε μια επιστολή που και αυτή την έχω στα χέρια μου στις 7 Ιουνίου. Και λέει κάτι περισσότερο στην τελευταία παράγραφο της επιστολής. Ο κύριος Μωράης αναφέρθη στο άρθρο 5, στον κανονισμό 539 του 2001 το άρθρο μάλλον 265 της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπε στον κύριο Αβραμόπουλο τα εξή. Κύριε Αβραμόπουλε, εξ ονόματος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι βάσει του άρθρου 265 των συνθήκων θα μπορούσε να υπάρξει ε, προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να υποχρεωθεί η Κομισιόν να δράσει. Ωραία. Ε, αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μετά τη δεύτερη ανακοίνωση η Κομισιόν θα ακολουθήσει μια τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και άλλες ανακοινώσεις. Αυτό που είναι απόλυτα σαφές είναι ότι η Κομισιόν δεν τηρεί τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό 539 καθώς 2001. Αυτό είναι σαφές. Και εγώ σας λέω με κάθε ειλικρίνη αυτό που είπα και στο παρελθόν. Έχω μεγάλη αγάπη για τις Ηνωμένες Πολιτείες των... της Αμερικής. Δεν θέλω να υποχρεωθούν οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτείων να παίρνουν βίζες. Αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείες πρέπει να απαλλάξουν από την, υπο, από την ανάγκη βίζα στην Πολωνία, την Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Κύπρο και την Κροατία. Δεν έχει νόημα γιατί οι Καναδοί θεωρούν ότι κάποιοι είναι καλοί και κάποιοι είναι κακοί. Όχι. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. Και αν το κάνουν όπως υπονοούν σε θέματα ασφάλειας, όπως φαίνεται να υπονοείται, αυτό δεν έχει νόημα. Γιατί η Πολωνία είναι λιγότερο ασφαλής από τη Γαλλία ή η Βουλγαρία. Γιατί η, Βουλγαρία, γιατί η Κροατία είναι λιγότερο ασφαλής από την Ιταλία. Δεν, δεν, δεν βγάζει νόημα αυτό, δεν έχει κανένα νόημα. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να κατανοήσουμε είναι η αμοιβαιότητα και το μόνο το οποίο είναι αποδεκτό είναι να διατηρήσουμε την συνεργασία μεταξύ των δύο όχθων του Ατλαντικού αλλά σε συνθήκες αμοιβαιότητας. Κλείνω λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Μπορεί κάπως να υποβαθμίζω αυτά τα οποία θα μπορούσα να υποβαθμίσω αυτά τα οποία λέει η ανακοίνωση κομισιών. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Νίδη. Λέει η ανακοίνωση ότι στις 18 Ιουνίου, Ιουλίου έλαβε χώρα μια συνάντηση μεταξύ του κύριου Κέρι και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έγινε εκεί. Τι έγινε στις 18 λοιπόν Ιουλίου. Πέστε μας. Γιατί αλλιώς θα ανακαστώ να πω αυτό το οποίο σας λέω. Εμείς συγχαίρουμε τον εαυτό μας για την περίπτωση του Μπρουνέη. Έχουμε κάποιες ελπίδες που τρέφουμε για την περίπτωση του Καναδά, αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε μια πλήρη διπλωματική αποτυχία σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Mrs. Sippel, please, παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να τα πω λιγάκι απλώς, με απλό τρόπο και το απλούστερο θα ήταν να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Διάστεμέρα, ο οποίος με το δικό του τρόπο διπλωματικά και ευγενικά μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει και αυτό το οποίο μας συμβαίνει δεν είναι καθόλου διπλωματικό. Είναι ουσιαστικά ένα θεατρικό παιχνίδι. Είχαμε μια σαφή συμφωνία με τον Καναδά, είχαμε μια σαφή συμφωνία με τις ΗΠΑ σε κάποια στιγμή να φτάσουμε στην ελευθερία από προξενικές θεωρήσεις. Και μετά αυτές οι δύο χώρες δεν τήρησαν αυτά που είχαμε, είχαν υποσχεθεί. Και δεν βλέπω κανένα να εξανίσταται. Και δεν κάνουμε αυτό το οποίο ήταν η φυσιολογική διαδικασία και που είχαμε συμφωνήσει ότι θα γίνει και με τις δύο αυτές χώρες, δηλαδή να εκδοθεί μία κατεξουσιοδότηση πράξη από την Κομισιόν. Έπρεπε μέχρι κάποια χρονική στιγμή εφέτος να είχε αρθεί η ελευθερία προξενικών θεωρήσεων. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μια τρίτη και μια τέταρτη ανακοίνωση που θα ακολουθήσει από την Κομισιόν για όλα αυτά τα θέματα. Ενδεχομένω υπάρχουν και άλλε χώρε οι οποίε είναι έτοιμε να άρουν την ελευθερία από προξενικέ θεωρήσει για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα και εγώ δεν θέλω, όπω και ο κύριο Δία Δεμέρα, να άρω την ελευθερία από προξενικέ θεωρήσει για τι ΗΠΑ και τον Καναδά. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υποχρέωση που θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί από την Κομισιόν. Δεν μπορούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι αντικείμενο διάκρισης επειδή προέρχονται από μια συγκεκριμένη χώρα. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτών από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που του ζητούν να κάνουν αίτηση για προξενική θεώρηση ή για κάποιο άλλο λόγο, γιατί βρέθηκαν στη Συρία ή για τον Α ή τον Β λόγο λένε ότι αυτό είναι θέμα ασφάλειας, αλλά δεν υπάρχει παραμικρή εγγύηση ότι αυτό δεν θα συνεχίσει. Στην ε, περίπτωση λοιπόν που υπάρχει αμφιβολία, εδώ βλέπετε να είναι σε βάρος του κατηγορουμένου η αμφιβολία από τις αρχές των ΗΠΑ. Επομένως, δεν, αν δεν μπορούμε εμείς να βασιζόμαστε σε αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, γιατί συνάπτουμε συμφωνίες. Περιμένω από την Ευρωπαϊκή ε, ε, Κομισιόν μια πολύ πιο στεναρή στάση από αυτήν που έχει κρατήσει και νομίζω ότι και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να λύσουμε τα συμπεράσματα από αυτή τη στάση της Κομισιόν, εάν χρειαστεί. Ευχαριστούμε, Μπριγκίτ, για τα σχόλιά σας. Καλό είναι που αναφερθήκατε σε αυτό το ζήτημα, γιατί εγώ θέλω να το συζητήσουμε και στους συντονιστές. Οπότε καλό είναι που βρίσκεστε εδώ και που πήρατε το λόγο για το ζήτημα αυτό, γιατί θα συζητηθεί και με τους συντονιστές. Καλό ήταν λοιπόν που ήσασταν παρούσα για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε για τη σχόλιά σας. Αν δεν θέλει να μιλήσει κάποιο άλλο μέλος, θα ζητήσω τη Σλοβακική... Α, συγγνώμη. Ε, θέλετε να ακούσετε πρώτα τι έχει πει η Προεδρία και μετά να επανέλθετε, κύριε Λοπέζ, ε, ε, γιατί ίσως να υπεξεί κάποιο άλλο ζήτημα. Κύριε Σεβενάκη, παρακαλώ, πάρτε το λόγο. Είχατε πολλή δουλειά σήμερα, σας το είχα πει. Έτσι είναι οι Προεδρίες. Ευχαριστώ. Πράγματι με μεγάλη μου χαρά ε, απευθύνομαι στην Επιτροπή για δεύτερη φορά σήμερα. Ουσιαστικά ελάχιστα έχω να πω για το ζήτημα αυτό. Δεν έχει συζητηθεί επίσημα στο Συμβούλιο. Μετά από την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση της Κομισιόν, ήθελα να επαναλάβω ότι το Συμβούλιο έχει δεσμευθεί στον απότερο σκοπό τη επίτευξη πλήρου αμοιβαιότητα στο θέμα των θεωρήσεων για του Ευρωπαίου πολίτε. Δηλαδή, άρση του σημερινού καθεστώτο όπου ε, ορισμένοι πολίτε κάποιων κρατών μελών υποχρεούνται να έχουν θεώρηση για να ταξιδέψουν σε ορισμένε ε, τρίτε χώρε. Εάν ε, τεθεί από την Κομισιόν το θέμα της της πράξης, σας διαβεβαιώ ότι η Προεδρία θα το αντιμετωπίσει ως κατεπήγον το ζήτημα αυτό. Εδώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ας επιστρέψουμε τώρα στον κύριο Σιγητή την Κύριε Μέρα. Σύντομα κύριε Πρόεδρε, όπως πάντα έχετε, έχετε δίκιο. Πρέπει να ακούσουμε πρώτα το Συμβούλιο και αφού θα έχουμε ακούσει το Συμβούλιο, εγώ σημειώνω, σημειώνω κατά λέξη. Μας είπε ο Βλαδιμίρ, το Συμβούλιο έχει δεσμευτεί για πλήρη αμοιβαιότητα. Το σημείωσα και σας το λέω γιατί δεν θα ήθελα να χρειαστεί να το θυμίσω στη Σλοβακική Προεδρία. Είναι λοιπόν απολύτως δεσμευμένο για αμοιβαιότητα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. So indeed it was useful to, <laughs> to hear that, more useful than you thought. Uh, ε, πολύ χρήσιμο ήταν λοιπόν. Πιο χρήσιμο από ό,τι νομίζαμε. Ναι, παρακαλώ τώρα να απαντήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο λόγια από πλευρά μα. Εμεί συμμεριζόμαστε την ε, σύγχυση αυτή και εμεί είμαστε πλήρω ε, ε, προσιλωμένοι στην απόλυτη αμοιβαιότητα, αλλά το θέμα εδώ είναι όχι το αν θέλουμε να κάνουμε μια της πράξη, αλλά να προβούμε στην καλύτερη επιλογή ώστε να επιτύχουμε το στόχο που έχουμε. Αυτό είναι το οποίο διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Και με βάση τις διάφορες αυτές εκθέσεις θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε περαιτέρω για να μπορέσουμε έτσι πιο λεπτομερώς να σας εξηγήσουμε γιατί και πώς ε, αντιδρούμε και τη σημείο, την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχουμε πετύχει, πιστεύουμε ότι ο δρόμος που ακολουθούμε είναι ο καλύτερος. Και πάλι η ανακοίνωση δεν είναι μια εναλλακτική σε σχέση με την κατεξοδότηση πράξη. Απλώς θέλει να σας ενημερώσει και να σας δείξει ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνοψίζοντας να πω ότι ο κύριος Ντίας Δεμέρα παρουσιάζει πολύ εμπεριστατωμένα τη θέση της Επιτροπής, της Επιτροπής μας και ακριβώ με το σωστό τόνο που θέλαμε. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επαναλάβουμε όλα όσα ε, υπόθηκαν. Η κυρία Σίπελ ζήτησε ε, και ρώτησε την Κομισιόν να έχει μια πιο ισχυρή και σταθερή θέση. Πάντως, χωρίς να προκαταβάλω το τι θα πούν οι συντονιστές, γιατί πρέπει να πάμε στους συντονιστές, για μια ισχυρή διακομματική ε, πολιτική απάντηση, γιατί είναι διακομματικό το θέμα. Το αναφέραμε όταν πρόσφατα πήγαμε στη ΣΥΠΑ και το λέω αυτό και προς την Κομισιόν ότι θα πρέπει αυτό να θεωρήσει ότι είναι η θέση μας. Ήταν σκληρή η συζήτηση, αλλά πάντως θα πρέπει να το αναφέρουμε και πάλι. Χωρίς να προκαταβάλω λοιπόν το τι θα πούν και τι θα κάνουν οι συντονιστές, πιστεύω ότι θα πρέπει να κλιμακώσουμε την θέση μας. να στείλουμε μια επιστολή από πλευρά του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Δεν θέλω τώρα να πω τι θα είναι οι δράσει που θα κάνουμε, σε τι δράση θα προβούμε. Πάντω να κάνουμε κάτι, να ζητήσω από του συντονιστέ να εξετάσουν τα διάφορα επίπεδα ε, απάντηση που μπορούμε να δώσουμε. Ε, νομίζω λοιπόν πως η ανάλυση του κυρίου Δίας Δεμέρα είναι η σωστή. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε και μας παρουσιάσατε την θέση σας με πολιτισμένο τρόπο. Σας ευχαριστώ ε, συνάδελφοι και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 12. Στις 17 Ιουλίου ψηφίσαμε στην Επιτροπή την έκθεση για την παρουσίαση για την κατάσταση πρόοδου στις τριμερείς διαπραγματεύσεις με, για το ποιες χώρες θα πρέπει και οι πολίτες τους θα πρέπει να έχουν ε, θεωρήσεις ή όχι και όσον αφορά την αναθεώρηση του μηχανισμού ανάκλησης έχουμε εισαγητή τον κύριο Δεμέρα κατεβλήθησαν προσπάθειες για να προχωρήσουμε γρήγορα και γι' αυτό θέλω να δώσω και πάλι το λόγο στον ίδιο τον κύριο Δίας Δεμέρα να μας παρουσιάσει πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις αυτές και βεβαίω να δώσω το λόγο και σε οποιοδήποτε βουλευτή θελήσει μετά. Παρακαλώ. De ε, να σας ευχαριστήσω και πάλι, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς, θα πρέπει να ξαναμιλήσω για απόγνωση και σύγχυση. Το είπατε και το είπατε σωστά, ότι βιαζόμαστε και είναι επίγον να προχωρήσουμε με αυτό το θέμα, το οποίο συνδέεται με ζητήματα παράπλευρα μεγάλης σημασίας ε, όσον αφορά την πολιτική θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέεται με την Ουκρανία, τη Γεωργία, το Κωσυφοπαίδιο και με τη συμφωνία με την Τουρκία. Και αυτό που θα πω τώρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευθεί, να μεταφραστεί και ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς. Αλλά όταν αναφέρω την συμφωνία με την Τουρκία, αυτό που κάνουμε και γι' αυτό είναι και τόσο επίγουσα αυτή η έκθεση, είναι ότι λέμε στους Τούρκους στην ουσία προσοχή, αν δεν είσαι καλός στη δουλειά σου δεν θα σε αφήσω να παίζεις με, το, με τα κλειδιά και με την κλειδαριά. Αυτό τους λέμε όμως. Δηλαδή, σημαίνει δηλαδή στην ουσία έναν εκβιασμό ότι κάνουμε. Αυτό είναι αυτή η έκθεση όσον αφορά την συμφωνία με την Τουρκία. Όμως θέλω να σας ε, εξηγήσω περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Ιωτόβα, την κυρία Μακοφέη, τον Πέτρ Γερέκ, την Κριστίν Τεβιράκ, και την ε, κυρία Βαλέρο που, που πολύ σαφώς κατάλαβαν ποια είναι η θέση μας και την κράτησαν τη θεσμική θέση του Κοινοβουλίου για να προχωρήσουμε γρήγορα αυτή την έκθεση. Λοιπόν, στις 7 ε, Ιουλίου ψηφίσαμε την έκθεση στην ΛΥΠΕ και έλαβα τη δική σας έγκριση για να ξεκινήσω την διαπραγματευτική διαδικασία. Είχαμε πολλές ελπίδες γιατί επιτύχαμε ε, πλειοψηφία συνένεση της ομάδας εδώ στο Κοινοβούλιο. Όμως η απόγνωση και η σύγκρουση δεν γίνεται εδώ. Έρχεται από το Συμβούλιο, γιατί ακόμα μια φορά το Συμβούλιο δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και το επίγοντα χαρακτήρα που το ίδιο ζήτησε. Το ίδιο το Συμβούλιο ζήτησε να, επιγόντως να περάσει αυτό το θέμα. Συγκλήθηκε τριμερής διάλογος, κύριε Πρόεδρε, για να ενημερώσουμε την Κομισιόν και ε, τρεις τεχνικές συνεδριάσεις. Στόχο είχαμε να έχουμε μια διαθεσμική συμφωνία πριν από το καλοκαίρι. Δυστυχώ δεν τα καταφέραμε. Α, τώρα θέλω να σας εξηγήσω πού βρισκόμαστε, πράγμα το οποίο γνωρίζουν κάποιοι συνάδελφοι. Καταφέραμε να πετύχουμε μια συμφωνία σε, στα εξή σημεία. Πρώτον, δημόσια ασφάλεια. Δεύτερον, σύστημα εποπτείας. Τρίτον, δυνατότητα παρακολούθησης και μάλλον τροποποίησης από μια απλή πλειοψηφία των κρατών μελών και ε, έναρξη της ε, αναθεώρησης μέσα στο πλαίσιο της ε, Επιτροπής. Η δημόσια ασφάλεια, να σας εξηγήσω τι είναι, θα εκφραστούμε μέσω απειλών στη δημόσια ασφάλεια και αυτό θα συνοδεύεται από εκθέσεις από τις αρμόδιες αρχές. Όσον αφορά την εποπτεία αναφερόμαστε στο άρθρο 1 του κανονισμού καθώς και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στους διαλόγους απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Και επίσης έχουμε προβλέψει μια περίοδο 8 ετών για να γίνουν οι αλλαγές. Αυτά είναι σημεία συμφωνίας είναι η αρχή των διαδικασία με πρωτοβουλία της Κομισιόν. Υπάρχει μια πρόταση ε, ε, συμφωνίας ότι δηλαδή η Κομισιόν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Φαίνουμε κάποιο διακριτικό περιθώριο γιατί η Κομισιόν απλά πρέπει να κοινοποιήσει με βάση σοβαρά στοιχεία που θα αποτελέσουν τη βάση για να τεθεί σε ε, κίνηση ολόκληρο ο μηχανισμό. Και φυσικά ταυτόχρονα πρέπει να ενημερώνεται το κοινοβούλιο. Και τώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, σε αυτό είμαστε όλοι πολύ ε, δεσμευμένοι. Η Κομισιόν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη στη διάρκεια τη διαδικασία την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι τρίτε χώρε με τι οποίε ασχολούμαστε, αλλά και τη δυνατότητα πιθανή και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η ανάκληση και η αναστολή της χορήγησης θεωρήσεων στους πολίτες αυτών των τρίτων χωρών. Όπως βλέπετε έχουμε πετύχει συμφωνία, αλλά υπάρχουν ακόμα ζητήματα στα οποία έχουμε κολλήσει. Και αναφέρομαι στο Συμβούλιο. Και Μάλιστα θα το κατακρίνω, θα το επικρίνω. Είναι, έχει μπλοκαριστεί το σημείο της ε, δυνατότητας θέσης εφαρμογή αυτού του μηχανισμού από την ε, μια πλειοψηφία απλή κρατών και επίσης η δυνατότητα ε, αναστολής και η δυνατότητα σύνταξη εξοδότηση πράξεων. Αυτά τα θέματα δεν έχουν ε, βρει στη συνένεση. Για το Κοινοβούλιο είναι μια βασική αρχή όλα τα μέτρα που σημαίνουν σημαντική αλλαγή του κανονισμού να χρησιμοποιούνται μέσω του νομικού μηχανισμού της κατεξιδότησης πράξης. Αυτό ορίζει η συνθήκη της Λισαβόνας και πιο συγκεκριμένα η απόφαση του, ε, ε του, του ΔΕΚ του στις 25 Ιουλίου του 2015. Αυτό το γνωστοποιήσαμε στην ε, Σοβλακική Προεδρία και τη είπαμε ότι υπάρχουν τρεις δυνατότητες, τρία διαφορετικά κείμενα που δεν μας απομακρύνουν από τον κεντρικό μας στόχο, δηλαδή να βρούμε μια λύση. Όμως δυστυχώς Δεν ευρέθη συμφωνία. Ελπίζω ότι μετά τις ε, διακοπές θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε θεσμική συμφωνία, διοργανική συμφωνία. Και εξακολουθώ να ελπίζω ότι ως εισηγητής εξ ονόματος του Συμβουλίου θα μου δώσουν κάθερες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που σας ε, γνωστοποιώ. Τι θέλει να επιτύχει το Συμβούλιο με αυτή την πιθανή μονομερή ενεργοποίηση του μηχανισμού. Δεύτερον, για ποιε περιπτώσει θέλω να το χρησιμοποιήσει, γιατί μέσω εκτελεστικών πράξεων και όχι εξοδότηση πράξεων, τι χρόνο, θα, θα πότε μάλλον θα επιθυμούσαν να ε, αρχίσει να ισχύει αυτό το μέτρο και αν θα συντάσσονται εκθέσεις ε, ή όχι από πλευρά της Κομισιόν. Δεν, αναφο... δεν απαντούν, ε, να απαντήσουν. Εάν θέλουν να βρούμε διοργανική συμβιβαστική, θα πρέπει να απαντήσουν στα ερωτήματά μας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Είναι αυτή μια θεμελιώδης πτυχή και ε, χωρίς απαντήσεις δεν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να καθορίσουμε μια θέση και πολύ λιγότερο μια ασυμφωνία. Δεν έχουν την ε, δεν την, ε, μας λένε όλο ότι δεν έχουν την έγκριση να συζητήσουν άλλα πράγματα και να διαπραγματευτούν άλλα πράγματα. Ε, ας τι πάρουν. Εμείς έχουμε κάνει τη δουλειά μας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την δουλειά μας όπως πρέπει. Θα πρέπει λοιπόν από εδώ και μπρος να κάνει και το Συμβούλιο τη δική του δουλειά. Τίποτα περισσότερο δεν έχω να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δίας Δεμέρα. Κάποιο άλλο μέρος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Όχι. Όπως πάντα ήταν ε, πολύ πλήρης οι πληροφορίες που μας δώσετε. Ο κ. Παρμά θέλει να πει κάτι. Ο κ. Σαμενάκ. Θέλετε να κάνετε κάποια παρουσίαση όπως την τελευταία φορά. Δεν είναι απαραίτητο. Αν θέλετε να πείτε κάτι, συντομία. Ναι, ευχαριστώ. Μάλλον θα περιοριστώ σε μερικές ε, λίγες ε, παρατηρήσεις ε, για το θέμα αυτό. Θα σας κάνει εκπλήξη ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Σιγητή σε πολλά σημεία που ανέφερε. Το πρώτο είναι ότι φυσικά κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχαμε στις αρχές Ιουλίου η Προεδρία κατάλαβε ότι έχουμε καταλήξει σε πιθανή, πιθανό συμβασμό για πολλά ζητήματα που περιλαμβάνει η πρόταση. Επίσης συμφωνώ με τον εισηγητή όταν λέει ότι κάποια σημαντικά ζητήματα δεν έχουν ακόμα επιληθεί και ότι στα ζητήματα αυτά οι θέσει του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου φαίνεται να απέχουν αρκετά. Όσον αφορά τα σχέδια της Προεδρίας, εμείς έχουμε κάνει έρωση προς την Κορεπέρ στις 20 Ιουλίου όσον αφορά την έκβαση των τριμερών διαλόγων και θα συνεχίσουμε, σας διαβεβαιώ όλους, συνεχίζουμε τις εργασίες μας, ειδικότερα σε διμερές επίπεδο. ώστε να προσδιορίσουμε το καλύτερο μελλοντικό δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Η σχέση μεταξύ του αρχείου αυτού και του αρχείου της ε, απελευθέρωσης των θεωρήσεων με ορισμένε χώρες είναι κάτι που απασχολεί την Προεδρία και συγκλίνουμε τις απόψεις της Προεδρίας για την κατάσταση. Οπότε να σας διαβεβαιώσω ότι το γνωρίζουμε. Όσον αφορά τα άμεσα βήματα που προβλέπουμε για το άμεσο μέλλον όσον αφορά αυτό το θέμα σχεδιάζουμε να ε, παράσχουμε ένα σχέδιο κειμένου στον εισηγητή, το οποίο θα περιλαμβάνει ε, μια πιθανή συμφωνία ή τις πιθανές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί σε ορισμένα από τα ζητήματα και επίσης θα μεριμνήσουμε ώστε όλες οι απαντήσεις προς διάφορες ερωτήσεις που είναι σημαντικές για την Επιτροπή θα φτάσουν στα χέρια του εισηγητή σχετικά σύντομα. Τέλος, ε, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα μου ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο πέρα από την τρέχουσα κατάσταση και να επιτύχουμε πρόοδο όχι μόνο σε αυτό το αρχείο αλλά και στα αρχεία απελευθέρωσης από θεωρήσεις που σχετίζονται με αυτό. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αν ο κ. Δεμέρα δεν θέλει να επανέλθει. Ωραία, σύντομα, παρακαλώ. Μόνο. Ναι, εν συντομία, απλώς για λόγους αυροφροσύνης, διότι η αυροφροσύνη δεν είναι ασύμβατη με τη διαφωνία και με, την, με τον κατηγορηματικό χαρακτήρα της διαφωνίας μας, το Συμβούλιο θα πρέπει να θέσει και κάποια ημερομηνία που να συνοδεύει τις υποχρεώσεις που συνάπτει γιατί δεν έχει πει τίποτα για τις ημερομηνίε. Ένα σύντομο χρονικό διάστημα, τι σημαίνει χρονικό διάστημα. Θα θέλαμε να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη προθεσμία και τον κατάλογο των σημαντικών θεμάτων τα οποία αναφέρει στο κείμενο, να ξέρουμε το ταχύτερο δυνατό πότε θα γίνει κάτι τέτοιο αυτή τη βδομάδα, ίσως αύριο δεδομέ, αν γίνει δυνατόν αύριο, σας παρακαλώ, τίποτα, αλλά αυτά ήθελα να πω. Τα είπατε πολύ καλά κύριε Διαστημέρα, έχει καταγραφεί αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πλήρη παρουσίαση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η κατεξουσιοδότηση πράξη και βρισκόμαστε σε καλά χέρια μέσα ως εισηγητή. Θα έχουμε μια, επανα μια συζήτηση και πάλι αυτό το θέμα. Το ταχύτερο να δω για να δούμε πού βρισκόμαστε. Πρέπει να διτηρήσουμε την πίεση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και το προσωπικό για την συμμόρφωσή τους με αυτό το δύσκολο χρονοδιάγραμμα και την οδυνηρή επιστροφή στις 30 για να εξετάσουμε και τα δύο αυτά θέματα και μπορούμε τώρα περνάμε στα διάφορα το σημείο 13 εάν δεν υπάρχει κάποιο θέμα στα διάφορα η επόμενη συνεδρία σήμαση θα είναι 5 Σεπτεμβρίου στις 3 η ώρα και 8 Σεπτεμβρίου δεν διαβάζω τα, τα γραμματά σας στις 2 η ώρα. Όχι, στις 3, στις 2, στις 8 Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και κλείνει η συνεδρίασή μας.